Κύριε Πρόεδρε, με κυρίε και κύριοι, καλώς ορίζω την πολιτική προσήλωση και τη σκληρή δουλειά του Κοινοβουλίου, της Καθήλυνα αλλά και των γνωμοδοτικών επιτροπών, της εισηγήτριας κυρίας Λόπε Φοντανιέ για την ταχύτατη εκπαίδευση της εκθέσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάνατε ό,τι μπορούσατε για να ε, βοηθήσετε στην προαγωγή αυτού του νομοθετικού πακέτου στη διάρκεια της θητείας του τρέχοντος κοινοβουλίου. Χαίρομαι που συμμερίζεστε σε μεγάλο βαθμό τις φιλοδοξίες και τους στόχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πλάς, ένα ολοκληρωμένο ταμείο με ουσιαστικό, με σημαντικό προπολογισμό που θα συμπληρώσει τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και θα συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ένα ταμείο πιο, με πιο απλή διαχείριση, πιο ευέλικτη διαχείριση που θα εξασφαλίσει περισσότερη προστιθεμένη αξία για τον τελικό χρήστη, τον πολίτη δηλαδή, και πώς εκ τούτου θα ε, εξυγχρονίσει την αγορά εργασία, θα εξασφαλίσει καλέ συνθήκε υγειονομική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα απευθύνεται σε εκείνου που το χρειάζονται περισσότερο, θα συμβάλλει σε μια ε, γενικά ε, στεναρή κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά δηλαδή θα προσφέρει περισσότερη κοινωνική Ευρώπη το Ταμείο αυτό. Το Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει μια σειρά από τροπολογίες, εκ των οποίων πολλές ε, θεωρώ θετικές, γιατί προσθέτουν ε, ή τροποποιούν προς τη σωστή κατεύθυνση το κείμενο. Ε, υπάρχουν όμως κάποιες άλλες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την συμπερίληψη συγκεκριμένων ποσών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σε εθνικό επίπεδο, κατανομή δηλαδή σε εθνικό επίπεδο, και αυτό το αναφέρουν πολλέ τοπολογίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά θα ήθελα να σα πω εδώ ότι αυτό θα περιορίσει σημαντικά την ευελιξία του Ταμείου. Και έτσι τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν να ανταποκρίνονται στι εξελισσόμενε κοινωνικέ ανάγκε, κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα θα συμβεί. Και δεν θα έχουν και τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα θέματα που ενδεχομένω αντιμετωπίζει ένα κράτο μέλο ή κάποια κράτη-μέλη και τα οποία εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις συγκεκριμένε τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την εργασία και την κοινωνική καινοτομία. Η πρότασή μας στόχο έχει να συνδέσει τα σημεία αυτά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με ικανοποίηση σημειών, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει τη συγχώνευση των ταμείων, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά πως είναι αναγκαία η ευελιξία. Έτσι λοιπόν συγκεκριμένα ποσοστά που θα μπορούσαν να επανεισαχθούν ε, πάλι θα έπληταν την ευελιξία του Ταμείου. Δεν θα επέτρεπαν δηλαδή την ανταπόκριση, την αντίδραση σε νέε προκλήσει. Το Κοινοβούλιο και η Ιδιαίτερη Επιτροπή ΕΝΒΙ επίση προτείνουν σημαντικέ ε, τροπολογίε στο τμήμα που αφορά την υγεία του Ταμείου. Ωστόσο, βλέποντας βεβαίως ότι θέλουν ε, ιδιαίτερη έμφαση να δώσουν στο θέμα της υγείας και έτσι το πρόγραμμα για την υγεία να μείνουν χωριστό μέσον και το σέβομαι αυτό, αλλά η Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι ε, η συνοχή και η καλύτερη αποτελεσματικότητα μεταξύ των ταμείων και η συνοχή θα, έχουν καλύτερα, θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα στις δράσεις για την δημόσια υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα στηρίξουν τους ε, επαγγελματίες της υγείας αλλά και τις αρχές αρμόδιες για τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Έτσι λοιπόν μπορούμε να διαφυλάξουμε και συγκεκριμένο κλάδο για την υγεία που θα υποστηρίζει τις πολιτικές δημόσιας υγείας για την υλοποίηση του στόχου εξασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου ε, ε, δημόσιας υγείας. Ταυτόχρονα όμως θα μπορούμε να εξασφαλίζουμε πως σε κάθε τομέα δημοσίων ε, ε, κοινωνικών δαπανών θα περιλαμβάνεται και ένας κλάδος υγείας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και είμαι στη θέση σας τώρα για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει η συζήτηση. Επιτροπή Προϋπολογισμών. Κλονέκ Μοχά. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε εδώ να κάνουμε ένα κανονισμό που μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία για σωστά, δίκαια, αποτελεσματικά εργαλεία για την κοινωνική Ευρώπη που εμείς σοσιαλιστές και δημοκράτες ζητούμε εδώ και χρόνια. Η έκθεση και η Επιτροπή των Προπολογισμών βεβαίω υποστηρίζει την καλή αυτή έκθεση. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω τις εξής τρεις προτεραιότητες καταρχάς η αναβάθμιση ενός ταμείου που θα απευθύνεται στις, ε, στους ε, λιγότερο προνομιούχους και η καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά πάνω απ' όλα η ενσωμάτωση της εγγύησης για τους νέους έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι τράπεζες τροφίμων επίσης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, την πολιτική, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τα ε, επιστηστικά προβλήματα. Και επίσης μια ισορροπία μεταξύ των ταμείων που έτσι συγχωνεύονται, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει μια ευελιξία ενώ θα μπορεί να υπάρξει μια ευελιξία. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρει στόχοι και θα πρέπει να αγωνιστούμε και σε πεδίο απασχόληση και επιτροπή περιβάλλοντο. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπράντο Πενιφέ, ο οποίο αγωνίστηκε πράγματι παρά τι αντιδράσει, αντιστάσει και ε, έντονε μερικέ φορέ ορισμένων πολιτικών δυνάμεων που θέλουν ε, μάλιστα να μα κάνουν να πιστέψουμε μερικέ φορέ ότι είναι προοδευτικέ. Πρέπει λοιπόν τώρα να προχωρήσει η πρόταση αυτή στο ε, Συμβούλιο έτσι ώστε να κλείσει το θέμα και να είναι ανοιχτή να είναι διαθέσιμο το ταμείο στους ε, περισσότερους δυνατούς πολίτες. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Τώρα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε μέχρι τις 11 ή 11 και κάτι το πολύ πολύ. Παρακαλώ. Ο κύριος ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προεπολογισμού είναι βαθύτατα πεπισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να συνεχίσει ε, ε, στο μέλλον να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και την απασχόληση και με τη συγχρηματοδότηση για μια πιο κοινωνική Ευρώπη εφαρμόζοντας τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων ε, στον ίδιο κανονισμό. Και σύμφωνα με αυτούς τους στόχους πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ θα πρέπει να υποστηρίζει και να αποσκοπεί σε συγκεκριμένους στόχους. Ο πρώτος είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ποιοτική και σταθερή δουλειά ε, να γίνεται σεβαστή η εργασιακή νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παντού ε, και τα δικαιώματα των ε, ανέργων, εκείνων που αναζητούν δουλειά, των μακροχρόνια ανέργων, προωθώντας την κοινωνική οικονομία ταυτόχρονα αλλά και την αυτοαπασχόληση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Βεσέτες Μπρέσο από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι και εγώ θα περιοριστώ σε ορισμένα ειδικά σημεία για την έκθεση που συντάξαμε ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να πω το προτινόμενο κείμενο της Επιτροπής με βάση το κείμενο του Κοινοβουλίου αναγνωρίζει καλύτερα τους ευεργετούμενους, τις περιφέρειες κλπ. Για να υπάρχει καλύτερη αποδοτικότητα του κανονισμού και το ΕΚΤ-ΣΥΝ να λάβει υπόψη την περιφερειακή συνοχή. Επίσης χαίρομαι για τις προθέσεις της Επιτρόπου να απλουστεύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και να υπάρχει συνέργεια μεταξύ ΕΚΤ και άλλων ταμείων. Αυτό είναι παράγοντας βελτίωσης. Τέλος, η πρόταση της Επιτροπής ορίζει ε, τη διασύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ΕΚΤ θα πρέπει όμως να υπάρχει και ευελιξία ε, μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης εθνικής και περιφερειακής ε, γιατί χρειάζονται επενδύσεις ορίζοντας καλύτερα την πολιτική συνοχής και ευρωπαϊκού εξαμήνου έτσι ώστε το τελευταίο να έχει μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο ρόλο. Σας ευχαριστώ η κυρία Κάμερβερτ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την ε, συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα δικαιοσύνη όμω, διότι εξαρτάται πάνω απ' όλα η εκπαίδευση από το πορτοφόλι των, ε, της οικογένειας των γονιών. Το αγαπητό κατά τα άλλα πρόγραμμα Εράσμους ακριβώς αυτό θέλει να αντιμετωπίσει και γι' αυτό η ανάπτυξη του προγράμματος Εράσμους θέλουμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον να συνοδεύει την ε, υποστήριξη που προσφέρει το ESF ε, και να υπάρχει μια, ένα σχετισμός μεταξύ των δύο η κινητικότητα που μπορεί να προσφερθεί ε, και να αποτελέσει σημαντική εμπειρία για τους ε, νέους, για τους μαθητές και μαθητευόμενους, μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό ε, όφελος και διαβατήριο για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν νομίζουμε ότι μπορούν να έχουν χάρη σε αυτό πολύ σημαντική εμπειρία, όφελος και επιτυχία επαγγελματική στο μέλλον. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή και να δώσουν κύρια προτεραιότητα, πρωταρχική προτεραιότητα στα θέματα της εκπαίδευσης από εδώ και μπρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ όλους τους ομιλητές να περιορίζονται αυστηρά στο χρόνο που τους έχει χορηγηθεί. Παρατηρώ ότι οι συνάδελφοι των Σοσιαλιστών Δημοκρατών ξεπερνούν περισσότερο από ό,τι κάποιοι άλλοι. Το χρονομιλία του ο κύριος Χρυσόγονος, παρακαλώ έχει το λόγο, δεν τον βλέπω όμως στην αίθουσα. Και παρακαλώ τον κύριο Πόστ, την κυρία Πόστ να λάβει το λόγο. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, στόχος μας είναι να γίνει ένα εργαλείο το οποίο θα επιτρέψει την ε, εξέλιξη και την ε, ενίσχυση των πολιτών. Θα πρέπει να είναι ανοιχτό στο δυνατόν, επιβάλλει στο δυνατόν λιγότερε διακρίσει, θα πρέπει να εξασφαλίζονται καλύτερε προοπτικέ ε, διαβίωση για όλου και ζωή για όλου στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει οι διακρίσει και ο αποκλεισμό να καταργηθούν. Οι κοινέ αξίε των συνθήκων μας πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει λοιπόν χάρη στο ταμείο αυτό να εξασφαλίσουμε μια κοινωνία βιώσιμη μια κοινωνία στην οποία εμείς ήδη έχουμε προσιλωθεί με, την, ε, με το θεματολόγιο 2020 για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κυρία Λόπες Φοντανιέ, αλλά και τον Πράτο Μποναφέ για την εξαιρετική συνεργασία στις ε, συνεδριάσεις των σκιωδών. Και τήρησα και το χρόνο μου. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωράγια. Ε, όντως, τήρησες το χρόνο σου. Από την ε, Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών, η κυρία Κοσλόφσκα Ρέιεβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αξιότιμοι βουλευτές. Καταρχάς θα ήθελα να ε, συγχαρώ την εισηγήτρια και τους κοιόδη εισηγητές για το έργο του. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει στόχο την εκρίζωση της φτώχειας, ε, την προώθηση της κινητικότητας Όλα αυτά τα γνωρίζουμε εμείς. Και στην Επιτροπή Γυναικών κάναμε τροπολογίες με στόχο να αρθούν οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα ίδια προβλήματα έχουν διαφορετικά αίτια για τους άνδρες και τις γυναίκες. Δεν οφείλονται στους ίδιους λόγους ας πούμε, οι γυναίκες, γιατί χάνουν τη δουλειά τους ή είναι εκτός ε, ε, εργασίας, ε, διότι δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές φύλαξης των παιδιών. Για τους άνδρες είναι άλλοι οι λόγοι που τους οδηγούν εκτός εργασίας. Μπορεί να είναι προβλήματα υγείας. Άρα ε, θα πρέπει να έχουμε προγράμματα ε, που να προωθούν τη φύλαξη των παιδιών για τις γυναίκες και για τους άνδρες προγράμματα ε, προαγωγής της υγείας τους και συμβουλές για το πώς να προσέχουν την υγεία τους. Αυτό θα πρέπει να σπάσει και οι διακρίσεις έτσι ώστε τα γυναικεία δικαιώματα να είναι πιο παρόντα και εγγυημένα. Ο κύριος Κάζα τώρα από το ΕΛΚ παρακαλώ σκεφτείτε και το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μια κοινωνική ένωση. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερες, περισσότερες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση μας και οι προτάσεις μας να βασίζονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Ιδιαίτερα όταν πλήττονται διοδρομίες και εργασία των Ευρωπαίων πολιτών. Το νέο ΕΚΤ θα επενδύσει στους Ευρωπαίους πολίτες, θα βοηθήσει τους πολίτες στην εξέβρεση νέας εργασίας και θα προωθήσει μια μεγαλύτερη επένδυση, μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό το βασικό μέλημα. Δηλαδή θα χτίσουμε πάνω στις επιτυχίες μας και θα ενισχύσουμε γιατί θα έχουμε τέσσερα ταμεία κάτω από το ίδιο φάσμα. Νομίζω ότι η κοινωνική συνοχή όλο ένα και θα διευρύνεται, θα υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και θα ενισχύσουμε εν γέννη τον κοινωνικό τομέα, όπως ισχύει στην πρόταση που έχουμε ενώπιον ο έχει το λόγο, ο κ. Ευχαριστώ την ε, κυρία Φοντανιέ για την εξαιρετική εργασία. Θέλουμε ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων να οδηγήσει σε νέους πόρους που να είναι χρήσιμοι για τους Ευρωπαίους πολίτες. Εγώ συνεισέφερα με τις τροπολογίες μου για να ενισχύσουμε το κείμενο της Επιτροπής για την ε, κατάρτιση, εκπαίδευση, καταπολέμηση της φτώχειας και ούτω καθεξής. Θα έχουμε περισσότερους πόρους για το Ταμείο Εγγύησης των Νέων και μέσα στα πλαίσια της ψηφιοποίησης θα πρέπει να βοηθήσουμε τα φτωχά στρώματα και να εργαστούμε στην, ε, για την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Έτσι θα γίνονται, θα υπάρχει μάλλον και συνεισφορά ως προς το, το εισόδημα, το ελάχιστο εισόδημα που ισχύει στην Ιταλία. Και επίσης ε, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται προγράμματα ενσωμάτωσης, ενσωμάτωσης σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε εισαγάγει ένα νέο μέσο, την εγγύηση για τα παιδιά που θα επιτρέψει σε παιδιά τα οποία δυστυχώς δεν έχουν τα κατάλληλα για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση και σε μια αξιοπρεπή ζωή και διατροφή. Γνωρίζουμε ότι το κείμενό μας είναι φιλόδοξο, αλλά αντικατοπτρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου για την αξιοπρέπεια των πολιτών και τις κοινέ μας αξίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ζωηρό σας ενδιαφέρον. Ο κύριος Χότς έχει το λόγο από το ECR. Το ανανεωμένο ΕΚΤ ενισχύει την κοινωνική Ευρώπη, ενισχύει και τις υποδομές αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο έτσι ώστε οι πολίτες να λάβουν υπόψη την ψηφιοποίηση, την παγκοσμιοποίηση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη, να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ένα νέο πρότυπο κοινωνικής φροντίδας που θα λάβει υπόψη και τις δημογραφικές αλλαγές. Δεν είμαστε όμως απόλυτα σαφείς ως προς τις επενδύσεις για τους νέους ή τη βοήθεια ε, των ανθρώπων με αναπηρίες, την υποστήριξη των Ρωμά ή την υποστήριξη ΜΚΟ και ΜΜΕ. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας δεν θα πρέπει να αποτρέψουμε την διασυνοριακή συνεργασία. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και υπέρ των νέων. Ο κύριος Σελίμοβιτς από τους φιλελεύθερους ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και την Επιτροπή για αυτή την εξαιρετική εργασία. Μιλάμε, μιλάμε για την κοινωνική συνοχή, την βοήθεια των πολιτών και αύξηση της ανταγωνιστικότητας ανά την Ευρώπη. Το συζητήσαμε για μήνες και μιλήσαμε για ευθυγράμμιση των στόχων με τις ε, συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Χαίρομαι γιατί ενισχύσαμε την ε, κοινωνική οικονομία, την εκπαίδευση των παιδιών, την υγεία, την ψηφιοποίηση και ούτω καθεξής. Προωθήσαμε την απασχόληση των νέων. Φυσικά θα αντιμετωπίσουμε κρίσεις και στο μέλλον, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς επιτύχαμε να υποστηρίξουμε την μακροχρόνια ενσωμάτωση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής. Οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ, είτε σας αρέσει είτε όχι. Όποια και να είναι η πρότασή σας, οι χώρες υποδοχής θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και τα χρήματα για να ενσωματώσουν τους μετανάστες στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Και είμαι υπερήφανος ε, γιατί το επιτύχαμε αυτό. Επίσης, μεγαλύτερη υποστήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών και πρόσβαση για όλους στην εκπαίδευση. Φυσικά δεν θα επιτύχουμε θαύματα αλλά θα έχουμε μία καλύτερη και πιο δυνατή Ευρώπη για την, για την επόμενη θητεία. Ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Ράιντκε από τους Πράσινους έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί Επίτροπε ένα μεγάλο κοινωνικό χάσμα είναι από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το δημοψήφισμα για το Brexit έδειξε ότι υπάρχουν άνθρωποι και πολλοί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στον Βασίλειο, που φοβούνται ότι τα κοινωνικά τους προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται και εμείς οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε όχι φεύγοντας από την κοινότητα αλληλεγγύης που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κάνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δίκαιη κοινωνικά. Και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ε, μία από τις ψηφίδες που θα βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει ενεργειακή φτώχεια, η φτώχεια στη στέγαση, ε, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η μετάβαση, όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πρόταση αυτή έχει αποδείξει ότι είναι ε, έτοιμο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα της ανισότητας. Και τώρα έχει έρθει η ώρα να δείξει και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη την προθυμία τους, θέλουν να βάλουν σε κίνδυνο το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από την ΚΟΕ το λόγο έχει η κυρία Κούνεβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαπραγμάτευση για τα διαρθρωτικά δαμεία δεν μπορεί να γίνεται υπό το φόβο του οικογικού κόστους. Είτε θέλουμε κοινωνική Ευρώπη ή όχι. Ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνεται στο σύνολό του για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο και μειώνονται και οι δαπάνες για τα κοινωνικά ζητήματα. σε μια περίοδο που έχουμε νέες ανάγκες ένα πληθυσμό που γερνάει την νεολαία μας που δεν βρίσκει δουλειά το μεταναστευτικό τη φτώχεια που μαστίζει. η ευρώπη χρειάζεται επιτέλους να αποκτήσει ένα κοινωνικό πρόσωπο αλλιώς θα καταστραφεί από τη δίκαιη αγανάκτηση του κόσμου της. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένους στόχους για τα κοινωνικά ζητήματα και πρέπει οι στόχοι αυτοί να είναι το ίδιο δεσμευτικοί όπως οι οικονομικοί. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ε, και τώρα ερχόμαστε στο τέλος το τοποθετήσω από πλευράς πολιτικών ομάδων και ακολουθούν οι μεμονωμένοι ομιλητέ. Ο κύριος Χέτμαν έτοιμος να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ε, Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Με χαρά είδα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτή η συγχώνευση πολλών συμπληρωματικών μέσων ε, μπορεί να καταστήσει την στήριξη πιο αποτελεσματική ε, και πιο διαφανή. Τώρα έχουμε ένα ενιαίο στόχο με 11 επιμέρους στόχους που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την εισαγωγή στην αγορά εργασίας. Και ε, το Κοινοβούλιο θέλει να τονίσει το ρόλο των περιφερειών, διότι οι περιφερειές δεν είναι απλώς δικαιούχοι ή κάποιοι θεσμοί που διαχειρίζονται τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ, αλλά... Ε, ασχολούνται και περισσότερο με τους πολίτες. Στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, έχω τη χαρά να σας πω ότι ε, βρήκαμε ένα συμβασμό με τον οποίο μπόρεσαν να συμφωνήσουν οι περισσότερες πολιτικές ομάδες και ελπίζω να μπορέσουμε να τα διαπραγματευτούμε και με το Συμβούλιο έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να εγκριθεί το έγγραφο. Ευχαριστώ κυρία Γιον Χέριου. ευχαριστώ πρόεδρε. Η φτώχεια είναι το δηλητήριο στις χώρες μας. Στην Ευρώπη ένα στα τέσσερα παιδιά κινδυνεύει με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό είναι παιδιά τα οποία στη συνέχεια μεγαλώνουν, γίνονται έφηβοι και αργότερα ενήλικοι που κινδυνεύουν να μην μπορούν ποτέ να καλύψουν αυτό το κενό και αυτή την ε, καθυστέρηση που έχουν και στην ε, εργασία και στην υγεία και έχετε απέναντί σας μία υπερήφανη ε, σοσιαλδημοκράτη. Εμείς ε, είχαμε την πρωτοβουλία να φέρουμε στο Κοινοβούλιο την εγγύηση για τα παιδιά και το Κοινοβούλιο κατάφερε να απελευθερώσει 5,9 ε, δισεκατομμύρια για την ναι, υπόθεση αυτή. Αλλά ε, τώρα η παιδική φτώχεια ε, εξαπλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και Θα πρέπει να εκριζωθεί και βοηθάει πάρα πολύ συγκεκριμένη έκθεση προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Παλώμα Λόπεθ Μπερμέχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να αξιολογήσω θετικά την ύπαρξη την ίδια του Ταμείου αυτού και του στόχου του για να χρηματοδοτεί τις κοινωνικές πολιτικές και την απασχόληση. Πλην όμως αυτό το εργαλείο και το μέσο που μπορεί να είναι καλό χωράει βελτίωση, τουλάχιστον στα εξή σημεία. Πρώτον και βασικότερο, θα πρέπει να έχει περισσότερα χρήματα αφού έχουμε ρίξει τους Ευρωπαίους εργαζόμενους στη φτώχεια, αυξάνεται και το κοινωνικό κόστος και το εργοσιακό κόστος, πολύ περισσότερο. Δεύτερον, θα πρέπει οπωσδήποτε να ταξινομήσουμε, να ιεραρχήσουμε τα ε, προγράμματα προτεραιότητας, δεξιότητες, ε, πρόγραμμα για τους νέους κτλ. Γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνέργειες με άλλα ταμεία, βέβαια με εξαίρεση το ε, EU. Όλα αυτά δεν πρόκειται να φτάσουν για να λυθούν όμως τα διαρθωτικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν τερματίσουμε ε, αυτό το κορσέ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σοφία Ριμπέιρο. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Συνάδελφοι, πιστεύω το ΕΚΤ ΣΥΝ να ενισχύσει τις προτεραιότητες του πυλώνα των ε, κοινωνικών ε, υποθέσεων και δικαιωμάτων. Θα πρέπει να είναι ένα απλουστευμένο πρόγραμμα ως προς την πρόσβαση σε αυτό και θα πρέπει να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να μην αποτελέσει ιδεολόγημα των κομμάτων. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζονται προγράμματα μεγαλύτερης ε, κοινωνικής συμμετοχής όπως η εγγύηση για τους νέους. Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιφέρειες που έχουν ε, ιδιαίτερες ανάγκες, που με οδηγεί και στο τελευταίο. Είμαστε η Ευρώπη των περιφερειών και θα πρέπει να άρουμε τα χάσματα που υπάρχουν ε, δίνοντας ε, διαφορετικές απαντήσεις για μια διαφορετική πραγματικότητα. Η κυρία Μπλινκεβιτσούτε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτό που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίσουμε τον υψηλό δίκτυ φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να χτίσουμε την κοινωνική Ευρώπη και να προωθήσουμε την απασχόληση καθώς και την ισότητα των δύο φύλων. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την φτώχεια των παιδιών και γι' αυτό να βρεθούν τα κατάλληλα μέτρα. Ε, το 1 τρίτον του ΕΚΤΣΙΝ θα πρέπει να προορίζεται στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γι' αυτό ζητούμε 6 δις ευρώ για την εγγύηση των παιδιών, για να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια στους ανηλίκους. Επίσης, ε, η συντάξει των γυναικών είναι κατά 40% χαμηλότερες από των ανδρών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα αντιστάθμισμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριος Δετιέ. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μόνο αυτό το οποίο μπορεί κανείς να ζήσει, να έχει την εμπειρία του, μπορεί να το θεωρήσει μακροπρόθεσμα καλό και θετικό. Έχουμε λοιπόν χρηματοδότηση προγραμμάτων στην Ευρώπη που βοηθούν τους ανθρώπους στην ε, καθημερινή τους ζωή. Ιδιαίτερα στις περιοχές που δεν έχουν τόσο καλή οικονομική ανάπτυξη, Φταίει συχνά το ερώτημα τι μας έχει προσφέρει η Ευρώπη. Το Κοινωνικό Ταμείο λοιπόν δίνει μια σωστή, μια αποφασιστική απάντηση. Η Ευρώπη είναι φτιαγμένη για τους ανθρώπους δίνει την κοινωνική εξασφάλιση, την ενσωμάτωση και πάλι στην κοινωνία, την υποστήριξη στην εργασία, την υποστήριξη του στην κοινωνική ζωή. Όλα αυτά τα προσφέρει το κοινωνικό ταμείο στην ε, ε, περίπτωση κλεισίματο επιχειρήσεων και μαζικών απολύσεων η Ευρώπη δεν αφήνει του ανθρώπου ε, μόνου του δεν του εγκαταλείπει ε, αγωνίζεται για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και γι' αυτό ζητούμε και τα παιδιά τα οποία πλήττονται από τη φτώχεια να έχουν τα βασικά δικαιώματα που είναι το δωρεάν σχολείο, τα δωρεάν σχολικά εγχειρίδια και την υποστήριξη ακόμα και για τη σχολική εκδρομή αν δεν μπορούν οι γονείς να τα προσφέρουν. Σας ευχαριστώ. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Η κυρία Ευλίν Ρέγκνερ έχει το λόγο. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χρειαζόμαστε χρήματα για να, για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων, για να δώσουμε στους νέους προοπτικές, για να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά στην Ευρώπη, να τους δώσουμε θέρμανση στο παιδικό δωμάτιο. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο, να έχει μια εγγύηση παιδική, να έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγη κατάλληλη και σωστή τροφή, διατροφή. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί και όχι να περικοπεί το ταμείο, το ESF+. Αυτό πρέπει να γίνει ώστε να μην περιοριστούμε μόνο στα ωραία λόγια. Εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδείξουμε ότι τα λόγια τα ωραία τα κάνουμε πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα τρία δευτερόλεπτα που μας δώσατε. Διαδικασία καρστία, κυρία Γεζογουέσικε. Ένα λεπτό. Το κλειδί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι η διαρκής κατάρτιση και η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Οι χρηματοδοτούμενες λοιπόν δραστηριότητες πρέπει να προσφέρουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες που είναι πράγματι ε, σημαντικές και απαραίτητες για την αγορά εργασίας, παραδείγματι ψηφιακή κατάρτιση. Έχουμε μια νέα ε, βιομηχανική επανάσταση, την ψηφιακή επανάσταση που απαιτεί αυτή την κατάρτιση που χρειάζομαστε ανθρώπους με καλύτερες δεξιότητες, νέους που θα μπορούν να προσαρμοστούν συνθήκες αγοράς εργασίας και άρα χρειάζονται ε, και τα ποσά εκείνα της χρηματοδότησης που θα επιτρέψουν την πρόβλεψη των εξελίξεων. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, τους εισηγητές για το Ταμείο και Πρέπει να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. για τους νέους που δεν είναι στο σχολείο, δεν εργάζονται ή δεν, έχουν, δεν είναι σε πρόγραμμα κατάρτισης, χρειάζεται ιδιαίτερη μέρη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ward, ένα λεπτό, χωρίς μικρόφωνο οι άνθρωποι με αναπηρίες, οι νέοι, νεαροί κατάδικοι ε, και άλλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστούν επιπλέον υποστήριξη γιατί θα χάσουμε 500 εκατομμύρια λίρες που προέρχονται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο, και φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε λοιπόν υπολογίσει ότι με την απώλεια και του ESF και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης οι υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες νέων θα χάσουν ε, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες λίρες το χρόνο όταν υλοποιηθεί το Brexit, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σημαντικά ποσά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα για τους νέους που έχουν πληγεί από την ε, λιτότητα. Από το 2010 που ανέλαβαν οι τόρεις, 710 εκατομμύρια λίρες αντιστοιχούν σε 710 εκατομμύρια λίρες αντιστοιχούν οι περικοπές ιδιαίτερα στις πιο φτωχές περιοχές όπως το Merseyside, η περιοχή μου, με 800 ε, με 800 νέους ανεργούς που θα χάνουν κάθε χρόνο την υποστήριξή τους την υποστήριξη που λαμβάνουν για επανακατάρτιση, αλλά και πολλούς άλλους που δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να, να εξασφαλίσουν νέες δυνατότητες για προσαρμογή στις δύσκολες συνθήκες της ζωής. Το Λίβερπουλ είχε ψηφίσει υπέρ. Ευχαριστώ σας διακόπτω γιατί έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Ο κύριος Μαριάς. Πρόεδρε, η παγκοσμιοποίηση, η λιτότητα, η βία, η δημοσιονομική προσαρμογή έχουν δημιουργήσει εκατομμύρια φτωχούς και ανέργους και είναι προφανές ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο πλας με τις δράσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβει μπορεί να κινηθεί σε διάφορα επίπεδα. πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσει την παιδική φτώχεια διότι η παιδική φτώχεια έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. να στηρίξει τους μακροχρόνια ανέργους να στηρίξει τους νέους μας οι οποίοι αναζητούν εργασία ταυτόχρονα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία κατάρτισης επιμόρφωσης για να μπορέσουν να σταθούν στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. επιπλέον τα άτομα με ειδικές ανάγκες νομίζω ότι και αυτοί χρειάζονται τη στήριξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου το οποίο μπορεί να απλώσει σε πολλά επίπεδα ακόμη και στο επίπεδο της ε, υγιεινής ε, των δράσεων που έχουν σχέση ε, με την απασχόληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πιμέντα Λόπες. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τους, τους απότερους στόχους του ΕΚΤΣΙΝ αλλά δεν πρέπει να υποκλίνεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στο πρόγραμμα της Επίτροπης που προωθεί και με το Invest EU. Ιδιαίτερα στην ε, Πορτογαλία βλέπουμε ότι οι εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ο τομέας της υγείας και της εκπαίδευσης δεν αναπτύσσεται. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις κοινωνικές προκλήσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας. Γιατί ε, έτσι μόνο θα έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικά στο ταμείο. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί τηρήσατε απόλυτα το ε, χρόνο σας. Η κυρία Σόιτροβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτός ο νέος κανονισμός για το κοινωνικό ταμείο θα οδηγήσει σε καλύτερη χρηματοδότηση, δεν θα υπάρχει πια επικάλυψη των διαφόρων ταμείων και έτσι θα έχουμε καλύτερη εφαρμογή του πλαισίου χρηματοδότησης. Θα υπάρχει λιγότερη, λιγότερος διοικητικός ε, φόρτος. Ε, Συμφωνώ με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο γιατί έτσι θα προσδώσουμε τους πόρους εκεί όπου υπάρχει καλύτερη αποδοτικότητα για να, αντιμετωπιστεί, να αντιμετωπιστούν και οι οικονομικές διαφοροποίησεις στα κράτη-μέλη. Καλύτερη λοιπόν ευελιξία, περισσότερη ευελιξία για καλύτερη χρήση των χρημάτων. Στην τσεχική δημοκρατία θα υποστηρίζουμε τις ομάδες των παιδιών που αντιμετωπίζουν μεγάλη φτώχεια. Κυρία Κονιέτσκα, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Είναι λυπηρό γιατί στις κοινωνίες μας υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. 100.000 βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης ένδυας. Ε, υπάρχουν πολλοί στην Τσεχική Δημοκρατία που αντιμετωπίζουν ε, και το φάσμα της ε, κατάσχεσης των περιουσιακών του στοιχείων. Έτσι ε, δημιουργείται και ένα φάσμα μεγάλων κινδύνων κοινωνικής επιβίωσης και χαίρομαι γιατί αυτό το ταμείο θα βοηθήσει τους ανθρώπους στην εκπαίδευση, η υγεία, δημόσιες υπηρεσίες, και κοινωνική συμμετοχή. Θα πρέπει να γίνονται περισσότερες επενδύσεις στους πολίτες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σεφάρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχανώ την κυρία Λόπε Φοντανιέ για την εξαιρετική της εργασία. Ε, πρόκειται για μία πολύ σημαντική ψηφίδα στις εργασίες μας και θα πρέπει να απασχολήσει περισσότερο. Μας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες υγείας μέσα στα πλαίσια της ε, πολιετής αντιμετώπισης Γι' αυτό το ΕΚΤΣΙΝ θα πρέπει να ασχοληθεί συνολικά με την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για 430 εκατομμύρια ευρώ συνολικά και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στην υγεία με μια βιώσιμη ανάπτυξη για να είμαστε πιο κοντά στον πολίτη και να υπάρχουν και κέντρα πληροφόρησης. Έτσι κανένας πολίτης δεν θα αφαιθεί εκτός αυτού του πλαισίου. Ε, Ρωμανά Τόμς, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν έχουμε υψηλό δίκτυ απασχόλησης και κοινωνική συμμετοχή, ιδιαίτερα ως προς τα χάσματα που υπάρχουν στην ψηφιοποίηση και την σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να είναι υψηλότερες. Το ΕΚΤΣΙΝ είναι ε, ένα επενδυτικό μέσο για το ανθρώπινο κεφάλαιο. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τους νέους μας και να θέσουμε μία ελάχιστη ποσοστιαία αναλογία συγχρηματοδότηση με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Η επίτροπο Τίσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Η συζήτηση αυτή έδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Και η έκθεσή σας θα αποτελέσει γερά θεμέλη για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Όπως πάντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαδραματίσει το ρόλο της ε, ως έντιμου διαμεσολαβητή στον τριμερή διάλογο. Ελπίζω να προχωρήσει και το Συμβούλιο από πλευράς του κατά τη Ρουμανική Προεδρία με στόχο να εγκριθεί εγκαίρος για τον επόμενο γύρο προγραμματισμού ε, η νομοθεσία αυτή, δυνατόν εντός του 19. Επενδύουμε στους ανθρώπους προάγουμε την ισότητα, τις ευρωπαϊκές αξίες, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική πρόοδο μέσω συγκεκριμένων δράσεων για να χειραφετηθούν οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, εργαζόμενοι άνεργοι, είτε έχουν γεννηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε έχουν γεννηθεί εκτός αυτής. Και μάλιστα από την παιδική ηλικία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ είναι ένα εργαλείο ε, για κοινωνική συνοχή και κοινωνική σύγκληση και μάλιστα είναι προβεβλημένο και ορατό για τους πολίτες. Ελπίζω όλοι οι συνομοθέτες και ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο να βοηθήσει έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκρίνεται στις θεμητές και εύλογες προσδοκίες ε, των πολιτών από το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά και για την ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών σας. Συγχαρητήρια σε όλους που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και ιδιαίτερα ε, στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η εισηγήτρια κυρία Λόπε Φοντανιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία του συναδέλφους και τη διαπραγμάτευση και βεβαίως να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Χρόνο δεν είχαμε πολύ, αλλά καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα γερό κείμενο ισόρροπο και αυτό το καταφέραμε χάρη στο γεγονός ότι όλοι είχαμε τον ίδιο στόχο, την κοινωνική βελτίωση της Ευρώπης στην Ευρώπη μάλλον και να αποφύγουμε κάποιες μαξιμαλιστικές θέσεις για να βρούμε όσο γίνεται μεγαλύτερο συμβιβασμό. Είμαι πεπισμένη ότι όλοι χρειάστηκε να κάνουμε ένα βήμα πίσω κάποια στιγμή, αλλά ε, ελπίζω, μάλλον είμαι πεπισμένη ότι θα βοηθήσει η συμφωνία αυτή στην οποία καταλήξαμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες όπου και αν ζουν για καλύτερη κοινωνική και οικονομική συνοχή ε, γράφεται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα και στο άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα ληφθούν υπόψη οι διάφορες ιδιαιτερότητες και διαφορετικές πραγματικότητες μεταξύ κρατών μελών αλλά και εντός των κρατών μελών όπως είναι ας πούμε η ε, απώλεια πληθυσμού από κάποια περιφέρεια. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτή είναι η βασική μας ε, ενασχόληση και το μέλημά μας να βελτιωθεί η ζωή τους. Και το δεύτερο ε, μήνυμα πηγαίνει προς το Συμβούλιο. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς τη δουλειά μας την κάναμε. Ε, ε, έδωσε καρπούς και αν εγκριθεί η έκθεση όπως ελπίζω είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Όσοι εισηγήτρια παρόλο που γνωρίζω ότι είναι δύσκολο ελπίζω κατά τη δερμανική Προεδρία εγκαίρως να λυθεί αυτό το θέμα για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και επιθυμώ και εύχομαι όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι να μπορέσει να ολοκληρωθεί η συζήτηση και η έκθεση αυτή κατά τη διάρκεια της παρούς κοινοβουλευτικής περίοδου. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λαπεφόντανιε. Και μπορούμε να σας συγχαρούμε πιστεύω ήδη. Ε, κλείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Περνούμε τώρα στο τελευταίο θέμα για απόψε. Μισή ώρα έχουμε προβλέψει ακόμα για τη συζήτηση. Έκθεση Πασκάλ Αριμόντ. Ειδικέ διατάξει που διέπουν το στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Ιντερέγκ. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Κοιτάξτε. Θα επιτρέψω ομιλητές να μιλήσουν στη διαδικασία αλλά που δεν έχουν ακόμα μιλήσει σε άλλες εκθέσεις και άλλο δεν σας παρακαλώ να ε, δείξετε κατανόηση και να το δεχτείτε αυτό. Ε, ε, είναι πολύ αργά και έχουμε τουλάχιστον 29 λεπτά ακόμα για τη συζήτηση. Για αυτή τη στιγμή έχουμε προγραμματίσει να τελειώσουμε στις 11 και 23 που είναι πολύ προχωρημένη ώρα. Το λόγο έχει ο εισηγητής. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα και την συζήτηση και την ψηφοφορία στην Βουλή των Κοινοτήτων. Απερίφθη λοιπόν η συμφωνία του Brexit. Το Brexit σημαίνει ταυτόχρονα και το τέλος του διασυνοριακής ε, κινητικότητας για τους εργαζομένους. Ακριβώς το θέτω από το Interreg. Και αυτό το πρόγραμμα Interreg, μπορώ να το πω από προσωπική εμπειρία, χρόνια τώρα από το 99 που συστήθηκε έχει βοηθήσει ιδιαίτερα τις ε, ε, παραμεθόριες περιοχές να ε, ζήσουν, να αναπτυχθούν. Πρέπει λοιπόν ό,τι εμπόδια υπάρχουν, ό,τι σύνορα υπάρχουν ακόμη και στο μυαλό των ανθρώπων να αποδιαρθρωθούν, να απαλληφθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και συμβολική το Interreg και γι' αυτό θέλω ιδιαίτερα να προχωρήσει το θέμα αυτό ε, 946 ήταν οι τροπολογίε οι κατέθηκαν, 46 οι συμβαστικές οι οποίες καταλήξαμε και εγκρίναμε στην Επιτροπή μας. Ομόφωνα υποστήριξαν το κείμενο όλες οι πολιτικές ομάδες και νομίζω αυτό ήταν και το χαρακτηριστικό. Στόχος μας ήταν ε, να μην είναι ε, αδιέξοδα οι περιοχές των συνόρων, να είναι ένα σημείο μετάβασης. Και πιστεύω ότι μπορούμε, μπορούμε να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστέλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 8,4 δισεκατομμύρια για την υπόλοιπη προγραμματική περίοδο χρειάζονται. Ο προπολογισμό που ξέρω βεβαίω ότι θα ε, παγιωθεί στη συνέχεια στι ε, συνομιλίε ε, και διαπραγματεύσει για το πολιετέ ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει αυτά τα 11,1 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, η διαπεριφερειακή, η διασυνοριακή, χωρίς περιορισμούς, χωρίς περικοπές. Πρόκειται για μια συνεργασία τεράστια σημασία και για την ίδια την Ευρώπη στο σύνολό της ε, ζωτική σημασία. Έτσι λοιπόν μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι περνούν τα σύνορα καθημερινά για να εργαστούν ε, που ουσιαστικά καταργούν τα σύνορα με τον τρόπο αυτό. Και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δούμε τι υπάρχει στην Ευρώπη, τι λειτουργεί καλά, τι δεν λειτουργεί καλά. Είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει τα πιλωτικά σχέδια, τα πιλωτικά έργα ε, με στόχο την καταργήση, την αντιμετώπιση των πολύ συγκεκριμένων προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν από τη μία πλευρά και την άλλη των ε, σύνορων και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η πρόταση με τα έργα ε, τα υπερσυνοριακά. Γι' αυτό χρειάστηκε να είναι πιο πολλά τα χρήματα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να μην χρειάζεται να αλλάξουν οι ε, φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται τα προγράμματα. Δεν υπάρχει λόγος εφόσον λειτουργούν ικανοποιητικά αυτά. Ε, δεν χρειάζεται. Ε, επίσης τα μικροπρογράμματα, αυτά που ονομάζουμε προγράμματα people to people από για τους πολίτες μεταξύ τους, ε, που έχουν μια πολύ συγκεκριμένη περιγραφή και προσδιορισμό στόχων, πρέπει να συνεχιστούν. Έχουμε νομίζω ότι ετυπώσει ένα κείμενο πολύ συγκεκριμένο πρακτικό δεν έχει, να κάνει, δεν έχει καμία σχέση με τον χρυσελεφάντινο πύργο των Βρυξελών όπως συχνά λέγεται. Μιλάει για αυτά καθημερινά προβλήματα. Έχει τη συνεργασία της Επιτροπής των Περιφερειών ε, έλεγχος ε, και γραφειοκρατία που θα πρέπει να υπάρχουν πάντα βεβαίως αλλά θα είναι περιορισμένοι και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει τώρα και πιστεύω ότι και οι προτάσει Ευρωπαϊκής Επιτροπής στείλουν προς την ορθή κατεύθυνση. Τα κριτήρια τα έχουμε ορίσει έτσι ώστε να είναι ε, κριτήρια που θα προετοιμάσουν ε, τα προγράμματα για το μέλλον, ε, παραδείγματι ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη κλιματική αλλαγή και άλλα ζητήματα έχουν ενσωματωθεί και μπορούν να καταστήσουν ένα ισχυρό σύμβολο αυτό το πρόγραμμα Interreg. Σκεφτείτε ότι ε, ήταν αναγκαίο για έναν, για έναν σκηνοθέτη που θέλει να κάνει μια ταινία για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος διακόπτη, ε, σας ευχαριστώ πολύ, έχει περάσει ο χρόνος σας και τώρα θα παρακαλέσω την κυρία Θεοχάρους, αλλά δεν τη βλέπω στην ένθουσα. Παρακαλώ λοιπόν την Επίτροπο Τίσεν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και πάλι μου δίνετε το λόγο. Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Άρμοντ και του και εισηγητές για την πολύ καλή έκθεση και την συνεχή υποστήριξη στην Ίντερεκ, την διεδαφική συνεργασία. Ιδιαίτερα η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, αξίζει συγχαρητηρίων για την ταχύτητα τη διεκπαιρέωση του φακέλου. Έχουμε πίεση χρόνου και έχει πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε έτοιμοι όταν ξεκινήσει η προσεχής προγραμματική περιοδο. Η Επιτροπή αισιοδοξεί ότι το Συμβούλιο θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνο ε, και κερδισμένο έδαφος αυτό το ε, πολύ σημαντικό θέμα και ότι θα εγκριθεί σύντομα. Η εδαφική συνοχή ή συνεργασία καλύτερα ε, όπως είπατε και εσείς, ε, αποτελεί το πολύ ισχυρό σύμβολο για την Ευρώπη. Ξεπερνούμε δηλαδή τα σύνορα, ξεπερνούμε τις αποστάσεις και υλοποιούμε κοινούς στόχους. Τα κύρια καινοτόμα στοιχεία είναι η αναδιατύπωση της αρχιτεκτονικής ώστε να αποκλειστούν επικαλύψεις και κατακαιρματισμό των έργων έτσι ώστε να είναι πολύ πιο στοχευμένες οι δράσεις του προγραμμάτος. Εδώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις ε, περιοχές λειτουργίες όπως θαλάσσιες λεκάνες αλλά ταυτόχρονα δίνονται και μέσα για την ε, διαφύλαξη και διατήρηση της ε, διασυνοριακής ή διαπεριφερειακής συνεργασίας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, παραδείγματι. Επίσης, μελλοντικά προγραμμάτα μπορούν να συνδέονται πολύ πιο ε, γερά με υφιστάμενα στρατηγικά πλαίσια και πολιτικές πρωτοβουλίες. Τέλος, απλούστευση του πλαισίου, ριζική απλούστευση, ώστε να δαπανώνται λιγότεροι πόροι στην διαχείριση και τον ε, έλεγχο και να στηριζόμαστε περισσότερο στα στόχους και την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως για την υποστήριξη που εκφράζεται προς την απλούστευση των στόχων αυτών και θα συνεργαστούμε μέσα σας βέβαια για την επίτευξή του. Τέλος, τα προγράμματα Interreg, διασυνοριακής συνεργασίας, εστιάζονται περισσότερο από πριν στην ε, συνεργασία μεταξύ θεσμικών αρχών για την επίλυση προβλημάτων ε, που έχουν να κάνουν με τα σύνορα και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Πάντα με απλούστευση, πάντα με διευκόλυνση της ε, διευρωπαϊκής συνεργασίας μπορούμε να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Επίτροπη, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, κύριο Κον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ είμαι ένα παιδί της Ευρωπεριφέρειας ε, ε, ε Ρήνου Μεύση που ζουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι ε, Βέλγοι, Γερμανοί, Ολλανδοί. Και είναι πολύ σημαντικό το Ιντερεκ. Ε, ρίχνουν τα σύνορα, συνεργάζονται πανεπιστήμια, συνεργάζονται επιχειρήσεις. Έρχονται οι άνθρωποι πιο κοντά ε, και πραγματικά το απολαμβάνουν και αυτό το στοιχείο της Ευρώπης. Και αυτό θέλουμε εμείς μια Ευρώπη που να ε, τη χαίρονται οι πολίτες και θέλουμε ε, μεγαλύτερη ενίσχυση των προγραμμάτων αυτών με περισσότερα χρήματα. Ε, δεν θέλουμε απλώς συνέχιση του έργου αυτού αλλά και ανάπτυξη του για να συνεχίζει η Ευρώπη να μεγαλώνει μαζί. Αλλά επειδή είμαι και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να μειωθεί το διοικητικό αυτό άχθος όταν η διοίκηση και η διαχείριση του προγράμματο χρειάζεται περισσότερο χρόνο από το ίδιο το πρόγραμμα, ε, δεν το χαίρεται τόσο πολύ ο κόσμο. Εμεί θέλουμε η Ευρώπη να είναι κάτι που να ενθουσιάζει και να αρέσει στου πολίτε. Γι' αυτό πρέπει να μεταξελιχθεί αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευση, κυρία Μίτση, παρακαλώ. President, l το χρηματοοικονομικό μέσο που χρησιμοποιείται εδώ έχει μεγάλη σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Είναι ύψης της σημασίας αν θέλουμε οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από το που προέρχονται. Ο πολιτισμός και η εκπαίδευση είναι ύψης της σημασίας αν θέλουμε να άρουμε τα σύνορα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη σωστή χρηματοδότηση. Θεωρώ ότι ο εισηγητής έχει επιτελέσει πολύ σημαντική εργασία, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε το τομέα της εκπαίδευσης, διότι έτσι βελτιώνεται και η ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποστέλουμε ένα μήνυμα. Όλοι είναι ίσοι, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Όποια γλώσσα χρησιμοποιούμε, όπου και αν βρισκόμαστε, χρειαζόμαστε ευκαιρίες. Ευχαριστούμε πολύ. Από το ΕΛΚΑ ο κύριος Βανίστελ Ρόι έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή Ερημών και την Επίτροπο Τέσεν. Πιστεύω ότι πραγματικά σήμερα φαίνεται ότι η διασυνοριακή συνεργασία δεν είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν, αλλά στο παρόν. Αν κοιτάξετε και μόνο τι γίνεται στη Βόρεια Ιρλανδία. Πρόσφατα είχαμε πάει εκεί με αντιπροσωπεία. Πώς συνεργάζονται τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και να πτήσουν νέα τεχνολογίες και στην ενέργεια αλλά και αλλού. Ε, και όλα αυτά τα εφαρμόζουν στην πράξη. Αυτό χρειάζονται οι παραμεθόριες περιοχές. Ε, είναι οι ουλές του παρελθόντος ε, ε, τα σύνορα και αυτές οι περιφέρειες. Και αυτό το βλέπουμε και αλλού. Και στη Σκωτία, ας πούμε, με τα προγράμματα Interreg, για παράδειγμα, πριν από 20 χρόνια βάλαν τα